Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτύου. Και τώρα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο 1 που είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως την οποία έχετε όλοι γιατί έχει μοιραστεί από τις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μία παρατήρηση μόνο να κάνουμε επ' αυτής. Ε, το σημείο 10 συγκεκριμένα Στις 27 Σεπτεμβρίου δόθηκε ε, μία σύσταση ε, σχετικά με, την, έναν κανονισμό ε, του Συμβουλίου που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Γενική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστοτικών ιδρυμάτων. Η εισηγήτρια ήταν η κυρία Τίσεν. Στο σημείο 10 λοιπόν θα πρέπει να ε, συζητήσουμε αύριο το πρωί για δύο εκθέσεις ε, σχετικές και θα έχουμε και την συνάντηση με τον Επίτροπο Σέρκοβιτς ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τις πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα το απόγευμα ε, θα έχουμε και την ε, έκθεση του συναδέλφου Τσαρκόφσκι. Θα ψηφιστεί αύριο. Και στις 5 θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συνεδριάσουμε μόνο με τους συντονιστές. Ah, sì, sì, certo. Allora, ho già una richiesta del Λοιπόν, ο συνάδελφο Άκνιου ε, θέλει να πει δύο λόγια σχετικά με την ημερήσια διάθεση, παρακαλώ. Είναι διαδικαστικό το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Ε, αέξω είπαμε ότι η συνεδρίαση είναι web streamed. Και την προηγούμενη φορά όμως είχαμε την ίδια ένδειξη, αλλά όταν ε, κοίταξα ε, για να δω την δικιά μου παρέμβαση και είδα ότι ε, όλη την ώρα που μίλαγα εγώ η κάμερα αντί να δείχνει εμένα έδειχνε μια χαριεστάτη νεαρή κυρία που καθόταν στο βάθος της αιθούσης. Ε, ε, βεβαίω. αυτό φαντάζομαι ότι μείωνε το εύρος των λόγων μου. γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι παραπονέθηκα στο, στη γραμματεία και μου είπε ότι σε κάποιες αίθουσες υπάρχουν κάποια νεκρά σημεία που δεν καλύπτονται από τις κάμερες. Ε, και γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ και ζητώ να μην με ξαναβάλετε σε ένα τέτοιο νεκρό σημείο. Ε, εδώ λοιπόν διάλεξα τη θέση μου και είναι ένα πολύ ζωντανό σημείο και εδώ θέλω να παραμείνω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, per me è un po' un problema, devo chiedere ai tecnici se quel posto dove lei si Βεβαίως, βεβαίως να καθίσετε εκεί έτσι ώστε να κινηματογραφήσετε κανονικά και με τον νόμο. Ε, αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό, λέει ο Πρόεδρος, ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Μας λέει, α ορίστε, η θέση που διαλέξατε είναι πάρα πολύ σωστή, κινηματογραφείτε σωστά η θέση σας, μου το επιβεβαίωσε και ο τεχνικός. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου, σημείο 2. Α, α, α, κι άλλο ζητάει το λόγο. Συγγνώμη, συνάδελφε Ντάφ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Βεβαίω θα πρέπει να συζητήσουμε και την έκθεση Kingold σχετικά με την τραπεζική αρχή για γνωμοδότηση. Τότε όμως, γιατί δεν συζητούμε την έκθεση Tyson για την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι δίδυμες αυτές οι εκθέσεις. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει ζητήσει το λόγο. Έχω και εγώ την ίδια παρατήρηση. Δεν έχουμε γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ. Δεν έχουμε γνωμοδότηση για την έκθεση Giggold. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό θέμα. Έχει περισσότερες ε, συνταγματικές έτσι, ε, επιπλοκές. Υπάρχουν συγκεκριμένα συνταγματικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με την αντίφαση ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, την Λυπή Ευρωπαϊκή Ένωση στην αυτή τη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε, έχουμε ακόμα χρόνο να ζητήσουμε τέτοια γνωμοδότηση. Η κυρία ε, Γιαννάκου, παρακαλώ. Euh, Κύριε Πρόεδρε, είχα την ε, εντύπωση ότι είχατε ξεκινήσει να συζητάτε την έκθεση ΝΤΑΦ, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι, δεν κατάλαβα καλά. Όχι, όχι, είμαστε στο πρώτο σημείο της ημερησίας εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, έγκριση της ίδιας. Εγώ είπα στην αρχή ότι στο σημείο 10 ήδη προεβλέπετο συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Τραπεζική Υπηρεσία. Εν τω μεταξύ όμως έχουμε και την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είπαμε ότι να τα συζητήσουμε αύριο και τα δύο. Ναι, ε, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί. Γουελτιέρη. Για να είμαστε σαφείς, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά θα, κάνουμε, ε, θα, ε, κάνουμε γνωμοδότηση, για την γνωμοδότηση και για την άλλη έκθεση, γιατί για την ώρα έχουμε έναν. Α, ο ίδιος λοιπόν, τώρα κατάλαβα, τώρα κατάλαβα, ο ίδιος θα ασχοληθεί και με την άλλη γνωμοδότηση. Δηλαδή, ο ίδιος εισηγητής. Ναι, ναι, αυτό εννοούσα, λέει και ο Πρόεδρος. Το είπα λίγο συμβιλικά, αλλά το ίδιο εννοούσα. Θα το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Ανακοινώσει eh, Ανακοινώσεις του Προέδρου. 18 και 19 Σεπτεμβρίου είχαμε επίσκεφτη στην ε, ε, Επιτροπή, της Επιτροπής μάλλον ε, στο Παρίσι. Ήταν μαζί μου ο Γουελτιέρη, ο Γκερέρο και συναντήσαμε κάποιους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου αλλά και του δικαστικού κόσμου καθώς επίσης και εκπροσώπους της ε, κοινωνίας των πολιτών στην Γαλλία κυρίως τον κύριο Σέρς ο οποίος ε, είναι και υπεύθυνος ε, για, πολιτικά, για ευρωπαϊκά θέματα και είχαμε και κάποιους άλλους εκπροσώπους, τον Σαλουί Ντεμπρέ, πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Φιλίπ Λεγκλής Κωστά, ο οποίος είναι σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για ευρωπαϊκά θέματα. Και βεβαίως συναντήσαμε και διανόμενους κτλ δεν ε, μπορέσαμε να ε, ε, πραγματοποιήσουμε τελικά την συνάντηση με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων γιατί μπλοκαριστήκαμε στην κίνηση και ήταν πολύ δυσάρεστο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να σας πω σχετικά με την επίσκεψή μας στο Παρίσι. Έχουμε τώρα το σημείο 3 και παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπή. θα συζητήσουμε το θέμα που αφορά τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες και το περιεχόμενο των εκθέσεων στο πλαίσιο τη διαδικασίας Έγκριση είχαμε ε, συζήτηση στα πλαίσια της Επιτροπής ε, των Προέδρων και διεφάνει ότι υπάρχουν έτσι διαφορετικοί κανόνες ε, για τις ψηφοφορίες στις διάφορες επιτροπές. Ο συνάδελφος Ταρκόφσκι λοιπόν την 19η Μαρτίου ορίστηκε εισηγητής για το θέμα αυτό και σήμερα ο ίδιος συνάδελφος έχει ένα έγγραφο εργασίας το οποίο τον καλώ να μας το παρουσιάσει. Yes. <coughs> Good afternoon. Καλησπέρα. The question which is before us is the question of clarifying rules of procedure on the Θέλαμε λοιπόν να, να συζητήσουμε τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες και το περιεχόμενο των εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης. Of those rules, because different committees behave in a different way, and recently we also had a problem when it came to the plea. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα καταλήξει η κατάσταση όταν φτάσουμε στην Ολομέλεια, δηλαδή τι θα πρεσβεύσει η Ολομέλεια σε, σε σχέση κιόλας με αυτό το οποίο έκανε με το άκτα. Acted with ACTA λέει κάνοντας λογοπαίγνιο στα αγγλικά ο μιλητή. και επομένω να δούμε τι προβλέπουν οι κανονισμοί σχετικά με αυτό. Να σα διαβάσω ε, αυτά τα τρία ερωτήσει. Πρώτα θα πρέπει οι τελείες παράγραφου να θεωρούν αποδεκτέ σε αυτό το σχέδιο του κειμένου και σχέση με το σχέδιο κειμένου που έχει προτείνει η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει οι τελεοπολίτες να θεωρούν αποδεκτέ στην ε, Ολομέλεια και στην Επιτροπή και ε, τι θα γίνει με την αρνητική ψήφο σε σχέση με την απόφαση θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ψήφος υπέρ ε, ή όχι. Αυτές, τα, αυτά τα ερωτήματα έχουν θέσει και το θέμα είναι το ότι ξέρετε όλοι τι έγινε όσον αφορά την διαδικασία αυτή. Θεώρησε ότι αυτό ήταν ένα τέχνασμα, ένα πυρηνικό όπλο για να, πει, ε, ε να χθεί το κοινοβούλιο να πει ένα ναι ή ένα όχι και με αυτό το πνεύμα διαπνέεται αυτή η διαδικασία αυτή εξ αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει βεβαίω και για μας το εξή θέμα. Θέλουμε να προτάξουμε την απόφασή μας ή θέλουμε πέραν αυτού να εξηγήσουμε γιατί ψηφίζουμε ναι ή γιατί ψηφίζουμε ου. Και όσον αφορά το κείμενο καθε αυτό, από τη διάταξη 81 προκύπτει αβίαστα ότι δεν έχουμε τίποτα τροπολογίες και δεν έχει φύγει το κείμενο της απόφασης όμως. Πάρα πολλές επιτροπές συμφωνούν σε αυτό το σχέδιο της ε, σύστασης. Έχουν μπει σε τουλικές παραγράφους που συνήθως αυτές οι παράγραφοι ξεκαθαρίζουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν προκειμένου το πρόβλημα είναι το εξή. Η πρακτική κάθε επιτροπή είναι διαφορετική. Κάποιε επιτροπέ υποβάλλουν ένα σχέδιο σύσταση και κάποιε άλλε όχι. Οπότε το θέμα που αναγύπτει είναι κατά πόσον ένα τέτοιο σχέδιο σύσταση είναι σαφές και αν επιδέχεται τροπολογία ή στην Ολομέλεια ή όχι. Εγώ έχω να σα πω τα εξή. Πρώτα πρώτα να διευκρινιστεί ποιο είναι το αληθε νόημα, ποια θα πρέπει να είναι η στάση του Κοινοβουλίου και επίση, όσον αφορά αυτέ οι ιτολικέ παραγράφου, αυτέ τι παραγράφου τέλο πάντων τη σύσταση, θα πρέπει να θεωρηθούν αποδεκτέ, παραδεκτέ, γιατί βοηθούν στο να διατυπωθεί θέση του Κοινοβουλίου και επίση θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να υποβληθούν τροπολογίες στην Ολομέλεια γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η απόφαση του να πούμε ναι ή όχι σε μια χώρα για να συνάψει σύμφωνο σύνδεση. Βεβαίω θα πρέπει να είναι η απάντηση ναι ή όχι, αλλά με ε, την σύσταση μπορούμε να πούμε γιατί λέμε ναι, γιατί λέμε όχι, μπορούμε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας και επίση να δούμε κατά πόσον υπάρχουν κάποιε έξτρα προποθέσει οι οποίες να, να, συνοδεύουν. Και επομένως θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, σίγουροι, κρυστάλλινοι σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Ναι λέμε ή όχι και αυτό είναι και το πνεύμα της συνθήκης και άρα δεν μπορούμε να παίζουμε. Από την άλλη μεριά όμως ε, τουλάχιστον θα πρέπει να, να, δούμε, να εξηγήσουμε ε, ποια είναι τα βασικά μας επιχειρήματα, τι έχει σημασία για μας, τι είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Ε, επομένως, στα ερωτήματα 1 και 2 θα πρέπει να απαντήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το περιθώριο ούτως ώστε να εκφράσουμε στην σύσταση τη γνώμη μας και να διευκρινίζουμε τι πρεσβεύουμε και επομένως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τροπολογίας. Η τρίτη ερώτηση όμως είναι πιο δύσκολη. Γιατί αυτό, διότι αν υπάρχει μια πρόταση συγκεκριμένης επιτροπής και συγκεντρώνει συνένεση και συμφωνεί και η Ολομέλεια όλα καλά. Όμως, όμως Ίσως το σενάριο να είναι το εξή, να γίνει απόρριψη της σύστασης της συγκεκριμένη επιτροπής. Και τι θα γίνει τότε, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτομάτως λέει ναι ή όχι το κοινοβούλιο και έτσι να διατυπώσει την αποψή της γιατί βέβαια έχει συζητηθεί στην στο, στο Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να δούμε και κάποια ενδιάμεση θέση. Δηλαδή, να έχουμε από τη μία μεριά αν υπάρχει τέλο πάντων διαφορά μεταξύ τη σύσταση επιτροπή και τη ψήφου τη Ολομελία, τότε να υπάρχει μια τρίτη εκδοχή να πούμε ότι απ, το Κοινοβούλιο ακόμα δεν αποφάσισε ή δώστε μας παράταση χρόνου. Και από αυτό επομένως θα πρέπει να είμαστε επίσης κρυστάλλινοι και ξεκάθαροι ότι εάν προταθεί μια τέτοια πράξη δεν συγκεντρώσει την Ολομέλεια να απορριφθεί. Ιδάλλως να θεωρηθεί στην αντίθετη περίπτωση ότι εγκρίνεται. Και αυτό να ισχύει αυτομάτω, δικαίως, ιδάλως ιδάλλως πρώτα-πρώτα αυτό που δημιουργούμε είναι νομικές περιπλοκές και δεύτερον αυτό μας δίνει μια τοποθέτηση πάρα πολύ ασαφή φλού. Και, και, και, σε σχέση με, με το άκτα, τι γίνεται. Έχουμε συνέπεια. Ε, Αλλιώ τα ανακατεύουμε όλα. Επομένω, με λίγα λόγια, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση μεταξύ μια πάρα πολύ στενή ερμηνεία της ε, συνθήκης να μπορούμε να πούμε ένα ναι ή ένα όχι με τις νέες ομάδες του Κοινοβουλίου γιατί θέλουμε υπορισμένες περιστάσεις να εξηγήσουμε τι αποφασίσαμε, γιατί το αποφασίσαμε. Και νομίζω ότι η συμβαστική λύση θα πρέπει να είναι στην σύσταση και στις τελικές παραγράφους ε, εάν, όταν έρθει η ώρα της τελικής ψηφοφορίας αυτό να είναι ξεκάθαρο, ένα ναι ή ένα όχι. Και άρα να προκύπτει ότι αν μία πρόταση δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία να θεωρείται απορριφθήσα. Ιδάλω να θεωρείται εγκριθήσα. Αυτά και τίποτα άλλο, διότι αν αρχίσουμε τους ελιγμούς θα υπάρξουν διάφορες ερμηνείες ε, θα θεωρηθεί ότι δεν αποφάσισε η αλφα η Β και μάλλον υπονομεύουμε και δεν αναδεικνύουμε το Κοινοβούλιο, στέλνουμε ένα αποδυναμωμένο, απονευρωμένο μήνυμα σε σχέση με τους ισχύοντες ε, κανόνες διαδικασίας, τον κανονισμό δηλαδή. Άρα ας συμφωνήσουμε σε αυτές τις παραγράφους, τις αιτιολογικές, ας συμφωνήσουμε και όσον αφορά τη διαδικασία, να μην υπάρξει αντιφάσεις ε, αν προστριβούντας των επιτροπών και όταν θεωρώ της ψηφοφορίας να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί, αλλιώς πάμε να μπλέξουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ε, τα επιχειρήματα του εισηγητού μου φαίνονται πολύ πιστικά. Γιατί είναι γεγονό ότι πρέπει να δώσουμε στο Κοινοβούλιο την δυνατότητα να, να επιχειρηματολογεί, να εξηγεί τη θέση του. Στη διαδικασία έγκρισης και όχι να έχει τη δυνατότητα να πει ναι ή όχι Ταυτοχρόνως όμως δεν θα πρέπει να υπονομευτεί και η σαφήνεια της τελικής ε, ψηφοφορίας. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια λογική συνέχεια βεβαίως. Άλλο είναι η λογική συνέχεια και άλλο είναι να υπάρξει ασάφεια ε, της έκβασης ε, της ψηφοφορίας. Και βάσει και των επιχειρημάτων λοιπόν που ακούσαμε από τον Σλάβ νομίζω ότι εύκολα μπορούμε να βρούμε λύση ε, στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Νταφ. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να επιτρέπουμε στο Κοινοβούλιο να εκφράζει την επιχειρηματολογία του για τις αποφάσεις του. Και μερικές φορές ήμασταν πολύ περιοριστικοί στην Ολομέλεια, στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν αφήσαμε να εκφραστεί το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις. σχετικά με τη χορήγηση έγκρισης. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση του Ραφάλ Τσαρκόφσκι και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το ναι ή όχι. Νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα προκύπτει εάν η συνθήκη και ο κανονισμός μας απαιτούν κάποιο κατόφλι για τη λήψη απόφασης. σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό το κατόφλι. Δηλαδή, αν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών, αλλά η απλή πλειοψηφία εκφράζεται αρνητικά ως προς τη σύσταση μιας επιτροπής, τι κάνουμε. Και φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην Ολομέλεια με νέα σύσταση από την Επιτροπή. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας στο σχέδιο έκθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ, Γκερέρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι σύντομος και θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε ο Ράφα, αλλά και με όσα είπε ο Ρομπέρτο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία που αφορά τόσο συγκεκριμένα ζητήματα, το Κοινοβούλιο επομένω να προβάλλεται ως ένα θεσμικό όργανο με τη δική του φωνή. Έτσι να το βλέπει ο κόσμος. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία τώρα μας προκύπτουν είναι ότι πολλές φορές, σε πολλές χώρες και για πολλού η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρείται ότι ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την Κομισιόν, με το, το Κοινοβούλιο. Δηλαδή από τη μία μεριά ε, μας, μας, μας μπερδεύουν και θεωρούμαστε ένα τμήμα της ουσίας αυτού του θέματος. Αλλά από την άλλη μεριά, πάρα πολύ συχνά, και νομίζω ότι όλοι το έχουν διαπιστώσει στη χώρα μας, το ότι υπάρχει το, το συνεχές ερώμενο ερώτημα. Τι λέει το Κοινοβούλιο, μα τι κάνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το α ή το β θέμα και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτή μας τη θέση. Ανεξάρτητα να τη διαμορφώσουμε και να την προβάλλουμε ακριβώς όπως προκύπτει από τις ε, συνθήκες και από την τελική ψηφοφορία όπως ε, προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Είτε πρόκειται περί σύμφωνης γνώμης, συνένεσης και επομένω να τοποθετηθούμε και να εξηγήσουμε και να μην αποφασίσουμε μηχανικά ή πίνα απλώ πατώντα το κουμπί τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ταρκόφσκι, νομίζω ότι ε, πρέπει να πω το εξή. Υπάρχει συνένεση από ό,τι καταλαβαίνω ε, στο να προσθεθεί στο ναι ή στο όχι μια αιτιολόγηση ε, και η αιτιολόγηση αυτή δεν έχω καταλάβει εάν θα πρέπει να συνοδεύεται από, ψηφοφορία. Ένα άλλο σημείο που είναι σαφές είναι όταν ζητάμε ενισχυμένη πλειοψηφία, απαιτείται δηλαδή ενισχυμένη μπορεί να κλείσει το θέμα με ένα ναι ή όχι ανάλογα με τον αριθμό των ε, ψηφισάντων ή ε, ε, θα πρέπει να, να συζητηθεί ξανά το ζήτημα. Δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά αυτό. Κύριε Ταρκόφσκι, παρακαλώ. Thank you very much for your comments. I think that the chairman... Ευχαριστώ για όσα είπατε και νομίζω ότι τα συνόψε πολύ καλά ο Πρόεδρος γιατί ακριβώς επί των περισσότερων σημείων για τα περισσότερα προβλήματα επίσης συμφωνούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται ε, με το κατόφλι ε, και εάν δεν πληρούνται το κατόφλι θα να θεωρηθεί ότι δεν έχουμε απόφαση και ίσως θα πρέπει να πάει να αναπευθεί στην Επιτροπή το θέμα. Αλλά κοιτάξτε, για να είμαστε σαφείς, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Εάν το κατόφλι αυτό δεν συντρέχει, τότε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης για να δούμε ακριβώς τι ισχύει ως πρακτική στο Κοινοβούλιο. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα και όταν έρχεται η ώρα της τεχνικής απόφασης με ψηφοφορία αυτές θα πρέπει να μην επιδέχονται αμφισβήτηση συγγνώμη αλλά κατ' δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση αλλά σημαίνει αν δεν το φτάσουμε το πλοίο αυτό, τότε σημαίνει τι το αντίθετο της αποφάσεως. Απόρριψη δηλαδή. Αλλιώς κάθε φορά θα υπάρχει αμφισβήτηση. Αυτομάτως να σημαίνει απόρριψη. Επομένως, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα και πάλι ας ρίξουμε μια ματιά στην, πρακτική του Κοινοβουλίου. τα κάπως περί, περί, έπλεξε τα πράγματα σήμερα και αν θέλουμε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση ε, τότε ο κόσμος θα μπερδέψει ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε δεν θα ξέρει τι λέμε και τι κάνουμε. Άρα δεν έχουμε κατόφλι. Δεν ε, έχουμε απόρριψη σημαίνει αυτό. Τόσο απλό. Εντάξει. Θα ζητήσω λοιπόν από τον συνάδελφο Τακόφσκι ε, ε, στις επόμενε συνεδριάσεις μας να παρουσιάσει το σχέδιο της έκθεσής του για να το συζητήσουμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Σχετικά ε, με το, τις ρήτρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμοιβαία άμυνα και ελεγγύη πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις. Εισηγητής, ε, συντάκτης μάλλον της γνωμοδότησης ε, είναι ο κύριος ε, Νταφ. Την 12 ε, Ιουλίου του είχε ανατεθεί, το Σεπτέμβρη είχε κάνει μια πρώτη παρουσίαση ε, της γνωμοδότησης που αφορά στην ουσία τροποποιήσει επί της ε, έκθεσης Πάσκου. Έχουν υποβληθεί 25 τροπολογίες και μπορούμε να συζητήσουμε επί των τροπολογιών αυτών, τις οποίες μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο. Κύριε Νταφ, συνάδελφε, θέλετε το λόγο παρακαλώ. Um, Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι επίγον το θέμα αυτό. Διότι η Επιτροπή έχει υποσχεθεί ότι θα είναι έτοιμη, έτοιμο το σχέδιο απόφασής της για την οργάνωση μιας ρήτρας αλληλεγγύης μέχρι τα τέλη του έτους και για να μπορέσουμε να ασκήσουμε κάποια επιρροή από αυτού πρέπει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου να ε, πάρουμε κάποια απόφαση για το θέμα. Δεύτερον, όπως βλέπετε, στη σύνταξη των γνωμοδοτήσεών μου συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την αρχή του εισηγητού κυρίου Πάσκου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Προσπάθησα να ασχοληθώ με τα συνταγματικά θέματα ή τα συνταγματικά στοιχεία αυτών των θεμάτων τα οποία προκύπτουν στην έκθεση Πάσκου. Και αφήνω τα θέματα κατεύθυνσης της πολιτικής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παραδείγματος χάρη, προτείνω κάποιες ε, προτάσεις του κυρίου Γιάννης Πανουέβο που είναι πιο κατάλληλες ε, για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θεωρώ ότι είναι πιο κατάλληλε για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων από ότι για τη δική μα Επιτροπή. Επειδή είναι επίγον το θέμα, ως προς τη διαδικασία προτείνω να κάνουμε άμεσα τροπολογίες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να μην ακολουθήσουμε την συνήθεια διαδικασία που συντάσσουμε γνωμοδότηση. Τρίτον, προσπαθώ να παραμείνω πιστός στη συνθήκη και να το εξηγήσω και να το δικαιολογήσω όπου είναι απαραίτητο. Και νομίζω ότι πρέπει ε, να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουμε υπόψη και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεργάζεται με τον ΝΑΤΟ. Η πρώτη ψηφοφορία αύριο αφορά το άρθρο 42, παράγραφο 7. Ο κύριος Πάσκου την αποκαλεί ρήτρα αμοιβαία άμυνα. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν ε, διαβάσουμε επακριβώς τη συνθήκη, καλό θα ήταν να το περιγράψουμε ως ρήτρα αμοιβαία ε, αρρωγής. Έτσι περιγράφεται στη συνθήκη. Ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. και για την άμυνα έναντι εξωτερικών επιτιθεμένων υπεύθυνο των ΝΑΤΟ. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά πρακτικής συνεργασίας. μεταξύ κρατών και ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Επίσης θέλω να αποφύγουμε την επανάληψη που μερικές φορές είναι αναπόφευκτη. στη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων ε, που ε, είναι παρεμφερείς. Αυτά είχα ως σχόλια. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίσω να απαντήσω. Και αν έχετε ερωτήσεις για τον κατάλογο ψηφοφορίας που έχει μοιραστεί, νομίζω, ευχαρίσω να απαντήσω. Βλέπω ότι η κυρία Γιαννάκου ξαναζήτησε το λόγο βέβαια. Φυσικά σας τον δίνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια αυτά τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Καταρχήν ε, ο κύριος Ντάφ επέλεξε έναν ιδιότυπο τρόπο να υποβάλει την εκθεσή του μέσω τροπολογιών πολλές των οποίων έχει ήδη υποβάλει και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μάλλον στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Μάλιστα ορισμένες εξ αυτών, όπως είναι τα σημεία 9, 10, 11 και 15, στις παραγράφους 4, 5 και 9, έχουν ενταχθεί σε, τροπολογ... σε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες Άρα τι νόημα έχει να ψηφιστούν εδώ αφού ήδη τα ίδια πράγματα έχουν ενταχθεί σε συμβαστικές τροπολογίες ε, στην ε, Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Ε, η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι, την είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, ότι δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί, κατά τη γνώμη μου, το defense clause για να μπει assistance clause, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η συνθήκη στο άρθρο 42 μιλάει συνεχώς για κοινή αμυντική πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών και επίσης διότι πουθενά η συνθήκη δεν θέτει όρους σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για το τι μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ είναι γνωστές στις χώρες αυτές. Και η αμοιβαία συνεργασία που πρέπει να υπάρχει εξυπακούεται, δεν συζητείται. Όμως αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε, δεν κάνουμε μια συζήτηση απλώς για να επαναλάβουμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση για μια ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης και άμυνας που αφορά στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν όλο το δικαίωμα είτε ανήκουν στο ΝΑΤΟ είτε δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ να δημιουργήσουν τους δικούς τους θεσμούς. Με ποια λογική δηλαδή εδώ ε, γίνεται μια πρόταση η οποία στοχεύει στο να υπονομεύσει αυτό που προτείνεται μέσω της συνθήκης. Εγώ είμαι αρνητική στην τοποθέτηση του κυρίου Νταφ, στην κεντρική του τοποθέτηση, διότι στην ουσία κάτι που πρέπει να γίνει, κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει, κάτι που αποτελούσε επιθυμία και των μελών της συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης και υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις και στην συνταγματική συνθήκη που ψηφίστηκε από πολλά κοινοβούλια και εν συνεχεία στη συνθήκη της Λισαβόνας προσπαθούμε να το βάλουμε σε μέτρα άλλων συμφωνιών και ε, συμμαχιών που υπάρχουν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο κύριε Πρόεδρε. Και ούτε είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε εδώ ότι ε, δεν αναφέρεται μέσα στη συνθήκη ε, η κοινή άμυνα. Το άρθρο 42 σε πάρα πολλές παραγράφους, στην 1, στη 2, στην 3, στην 4 και εν συνεχεία στην 5 και κυρίως στην 7 ξεκαθαρίζει ότι εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία πρέπει να αναλυθεί και που περιλαμβάνει βεβαίως και την μείωση των, του κόστους των εξοπλισμών και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Άμυνας και την ε, προσπάθεια στην παραγωγή όπλων ε, να υπάρξει ε, καλύτερος συντονισμός και όλα όσα μπορούν να γίνουν από μια ένωση που έχει δική της νομική προσωπικότητα. Αυτό νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί στην έκθεση του κυρίου Ντάφ. Η Ένωση έχει δική της νομική προσωπικότητα, κύριε Ντάφ. Και δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να θέσουμε την Ένωση υπό συνθήκες και συμμαχίες που έχουν υπογράψει κράτη-μέλη της με τρίτους αυτά τα κράτη-μέλη πάντοτε θα τηρούν τις συμφωνίες που έχουν κάνει και σε αυτό που θα φτιάξουμε θα περιλαμβάνονται και τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν σε άλλες συμμαχίες. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα ούτε η έκθεση που κάνατε εσείς, ούτε η έκθεση που έκανε ο κύριος Πασκούχαν με την ώρα μας. Επομένως θέλω να πω ότι είμαι τελείως αντίθετη με τη βασική αρχή η οποία εκφράζεται στην έκθεση του κυρίου Νταφ μέσω των τροπολογιών του αλλά και μέσω των τροπολογιών που έχει υποβάλει στην ε, Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας διότι απλώς στοχεύουν να εξαφανίσουν το νόημα που ε, έχει το άρθρο 42 της συνθήκης. Το άρθρο 42 είναι κατηγορηματικό, δεν αφήνει καμία αμφιβολία και δεν θέτει την προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει κάτω από την επιταγή οποιοδήποτε άλλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρόκειται για διαστρέβλωση πλήρη του άρθρου της συνθήκης όπως διατυπώνεται κύριε Πρόεδρε και βεβαίως σας σημειώνω και πάλι τα τέσσερα ε, σημεία τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε compromise ε, amendment, σε, σε συμβαστικές τροπολογίες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αφού έχουν μπει σε συμβαστικές τροπολογίες στην Υποεπιτροπή Άμυνας γιατί πρέπει να ξανάρθουν εδώ ως τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαννάκου, ο κύριος Γιάννετς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Να σας πω ότι η πολιτική ομάδα την οποία εκπροσωπώ συμφωνεί με το κοινωνικό πνεύμα των όσων είπε ο κύριος Νταφ. Και επίσης ότι ευθυγραμμιζόμαστε πάρα πολύ με τις ε, απόψεις ε, ουσίας του θέματος του κυρίου Πάσκου. Ίσως ε, πάντως από πλευρά ε, τεχνική, από πλευρά ε, διαδικαστική, αυτά τα οποία είπε ο κύριο Νταφ ε, και αυτά τα οποία είπε δηλαδή συγκεκριμένα όσο αφορά τι τροπολογίε, ίσω, ίσω, ίσω ορισμένου από εμά κάπω δημιούργησαν κάποια σύγχυση. Όμω, όμω, επί τη ουσία νομίζω ότι. το να άκουσα τέλο πάντων πιστεύω ότι συμφωνούμε. Και επίση νομίζω ότι υπάρχει υπάρχει αυτή η ρήτρα άμυνας και υπεράσπισης του ενός από τους άλλους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και επίσης υπάρχει αυτή η υποχρέωση αρρωγής, βοηθείας, συμπαράστασης και επομένως στο άρθρο 42 παράγραφος 7 διατυπώνονται αυτά που τα λέει αυτά ακριβώς και ο κύριος Ντάφη στην έκθεσή του και βλέπουμε ότι εδώ πέρα θέλουμε να ξευρωπαίσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή άμυνα, γιατί επί δεκαετίες ήταν και ακόμα είναι πάρα πολύ εξαιρετημένοι από το ΝΑΤΟ. Από τη ΣΥΠΑ δηλαδή, το Βρετανικό Σύμφωνο και οπότε ε, κάθε φορά που έχουμε τέτοια θέματα να μην λέμε τα ίδια. Δεν ε, θέλουμε με όλα αυτά να γίνουμε αντιαμερικανοί, να γίνουμε επικριτέ τον τον ΗΠΑ. Όμω θα πρέπει άποψη και διαπαντό η Ευρώπη να αναλάβει τι ευθύνε τη όσον αφορά την αμυνά τη, που θα πρέπει να αποκτήσει όσο γίνεται πιο ε, αυτόνομη και φυσικά ω χώρα με τη ΣΥΠΑ και με τον Όταν ω θεσμικό όργανο βεβαίω και συνεχιστεί η συνεργασία. Όμω αυτή η έκθεση ε, προσδίδει στοιχεία ποιοτικά, είναι ένα βήμα προ τα εμπρό. Ε, για αυτού του είδους την ε, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα δώσουμε στην άμυνα και ασφάλεια και σε αυτή την ε, έννοια της ταχείας απόκρισης. Οπότε, για αυτό το λόγο και έχουμε εδώ πέρα κατεβάσει και κάποιες τροπολογίες και εγώ ο εκεί στην 6 και στην 28 εκ μέρους πολιτικής ομάδας και λέμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε όσον αφορά την ε, διεθνή τρομοκρατία, όσον αφορά τα ανεξέλεγκτα κράτη, όσον αφορά και κάποιες ε, κρίσεις που σοβούν, που είναι τέλο πάντων ε, σε φάση που ακόμα συνεχίζονται και οπότε είτε εγκριθεί είτε όχι τέλο πάντων η θέση του κυρίου Νταφ έχουμε κάποιες απειλές, έχουμε κάποιους κινδύνους που δεν είναι του παραδοσιακού στερεωτικού χαρακτήρα. Είναι άλλου είδους αυτή η κίνδυνη και αυτές οι απειλές. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά νομίζουμε ότι σε αυτό το πολιτικό και νομικό έγγραφο το οποίο τώρα καλούμεθα να εγκρίνουμε όλα αυτά αποτυπώνονται. Οπότε και γι' αυτό και ελπίζω ότι αύριο θα τα βρούμε με τον εισηγητή και όλα θα πάνε καλά όταν έρθει η ώρα της, ψήφισης των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ, Λεπρόεδρος, ο επόμενος συνάδελφος τώρα, ο Σάγνου. Και ποιος άλλος θέλει το λόγο? Ναι, ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ. Εσείς, κύριε Άγνιου. Thank you. It's quite clear that what lies behind these είναι σαφές ότι το πνεύμα το οποίο υποκρύπτουν αυτά τα εγγραφά είναι αυτό το οποίο θέλουν αυτοί που θέλουν την Ομοσπονδιακή Φεντελεστική Ευρώπη να φτιάξουν ένα στρατό ευρωπαϊκό. Αλλά πρώτα πρώτα, για να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται εδώ. Εδώ, η ΣΤΕΛ θέλει να έχει μια υποδομή για να δημιουργήσει, να συγκροτήσει τέτοιο στρατό και ο στόχος είναι αυτή, λέγεται εδώ δίθεν εισαγωγικά, η αμοιβαία αρρωγή, ενίσχυση προς τα κράτη-μέλη, όλα αυτά δικαιολογούνται από τις συνθήκες. Από την άλλη μεριά όμως από την άλλη μεριά, όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ είναι μεγάλο βήμα που δημιουργεί το του Στρατού. Δεύτερον, όσον αφορά του φεντρελιστέ, ε, ποιο είναι ο σκοπό αυτού του στρατού, για να απαντήσω το ερώτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε εξετάσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. το περισσότερο της οποίας αφορά το πώ θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί την εξωτερική πολιτική όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε και έχουμε τώρα ε, ε, νευριακή καταστάση, ένα Υπουργείο Εξωτερικών και από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το μεγάλο όραμα ε, το του κάπω εθροβάμων, την διπλωματική υπηρεσία την ονομάζουμε και πάμε έτσι να φτιάξουμε και μια πολιτική ασφάλειας και, και, και, και άμυνας. Όλα αυτά πάμε σε αυτά που είπε ο κύριο Κλάουζεβιτ. Τι είχε πει ο Κλάουζεβιτ, είχε πει ότι ο πόλεμο είναι συνέχεια τη πολιτική με άλλα μέσα. Είπε ο Κλάουζεβιτ. Και εάν έχουμε μια τέτοια κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, θα πρέπει κανεί να έχει το στρατό για να την ε, υποστηρίξει. Ιδάλω, αντίο σα. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε πώ θα έχουμε την πολιτική αυτή, πώ θα έχουμε τον στρατό, γιατί μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιο είναι ο εγγυητή τη ειρήνη, είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο το στηρίζουν οι ΗΠΑ και φυσικά και η δική μου χώρα το Εμμήνου Βασίλειο. Οπότε θα πρέπει οι φεντελιστέ να βρουν τον τρόπο να, φτιάξουν τέτοιε ένοπλε δυνάμει. Αυτέ εδώ πέρα είναι οι φιλοδοξίε. Από την άλλη μεριά όμω με τον ψοφοδέη συνήθι τρόπο, εδώ πέρα μακαρεύεται το κείμενο να λέει κάτι άλλο. Όμω θα πρέπει να, να, να, να ξεκάθαρο. Θα πρέπει να έχουμε ένα στρατηγείο σταθερό ευρωπαϊκό. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε στο να έχουμε κάποιε επιχειρήσει ευρωπαϊκέ. Και να γίνουν επιχειρήσει θα χρειάζεται ένα στρατό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εδώ πέρα ξεκάθαροι ότι υπάρχει μηδέν υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συγκρότηση ενό τέτοιου ευρωπαϊκού στρατού. Δεν υπάρχει καμία τέτοια εντολή όσον αφορά τον Βρετανικό λαό για τη συγκρότηση τέτοιου στρατού. Και ο Βρετανό βουλευτή που κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα ξέρει πολύ καλά και ξέρουμε πού πάνε όλα αυτά. Εάν οι φεντεραστέ τα καταφέρουν, τότε κάποια στιγμή θα κληθούν να, να υπηρετήσουν κάποιοι νέοι Βρετανοί και θα του έχει διαλέξει αυτή η ελίτα των Βρυξελών. Αυτό ο Φαν πάει και από, από τα εγκριτό και παρεδίστο από τον Περλεμόν και τελευταίο θα σα πω ότι τελικά ο χειρότερο εφιάλτη θα είναι όταν αναλάβει τα Ινία ε, των πυρηνικών δυνάμειών μα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των, των όσων έχει κανονίσει η Γαλλία και ε, θα, θα λέμε ότι θα, θα, το, το κουμπί, το κόκκινο θα καλύτερα να το πατήσει πιο σοφάν ρομπόι. Και βεβαίω θα πρέπει για τι εκλογέ του 2014 να δούμε πώ θα εκτεθεί το κοινοβούλιο. Μάντριο, εσύ από του δικού σου ψηφοφόρου, τι εντολή έχει για να προωθεί τέτοια πράγματα. Okay, thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Η συζήτηση αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, αφορά την πολιτική και την επιχειρησιακή διάσταση. Και συνήθως οι σειράξεις γίνονται χωρίς προκαταρκτική σκέψη. Συνήθως γίνονται μετά από μία ή δύο πολιτικές αποφάσεις. Και συνήθως οι συγκρούσει, εσφαλμένα βλέπονται ω κάτι το οποίο ξεκινάει με εχθροπραξίε. Αλλά πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίε, μπορεί να υπάρχει ένα ολόκληρο κατάλογο φραστικών ε, ε, συμβάντων ή ιστορικών διεκδικήσεων και απαιτήσεων. Το ερώτημα του ποια χώρα ξεκίνησε αυτή τη δράση μπορεί να μην είναι ίδια όπω ε, το ποια χώρα προκάλεσε την σύγκρουση η χώρα μου και άλλες χώρες ε, δεν θα θέλαν να μπουν σε σύγκρουση που δεν είναι δική τους υπετιότητα. Ε, μια σύγκρουση την οποία δεν, καταλαβαίνουμε, δεν θα καταλαβαίνουμε επαρκώς. Όταν προσλαμβάνουμε προσωπικό, τους ε, προσλαμβάνουμε χωρίς να θέλουμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή τους. Με πολύ μεγάλη προσοχή χειριζόμαστε τα βήματά μας. και βλέπω και ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη δυστυχία της Κύπρου. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ πριν από τόσα χρόνια και πόσοι αλληλεγγύη έχουμε δείξει στην Κύπρο για να απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή. Αν δείτε το 42-7, σαφώς ε, αυτό μπαίνει στον ορισμό της ένοπλης επίθεσης ε, στο ίδιο έδαφος ε, στην ίδια επικράτεια της χώρας. Η Τουρκία δεν υπέστη καν ακύρωση του καθεστώτος της συνδεδεμένης ε, χώρας. Ε, κάτι το οποίο, ε, με το οποίο διαφωνούν και το οποίο φέρνουν βαρέως και οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι βλέπουμε τις λέξεις της τροπολογίας 10 και βλέπουμε ότι λέει ενίσχυση της Ευρωπαϊκής, δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητας. Και στο 11 λέει η υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και στην τροπολογία 18 λέει μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρώπης μεταξύ των πολιτών ε, που θα πρέπει να απολαμβάνουν το ωφέλη της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Με τις ρήτρες αμοιβαίας ε, άμυνας και αλληλεγγύης νομίζω αυτό το νόημα που υπάρχει είναι το ίδιο με οτιδήποτε άλλο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ενιαία αγορά μέχρι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ε, ούτε στρατιωτικοί ε, στόχοι, ούτε δημοσιονομικό σύμφωνο είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι το να προχωρήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η σταδιακή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ε, μετά την ε, παρέμβαση και την γνωμοδότηση της τροπολογίας του Άντριου Νταφ θα ήθελα να μιλήσω για το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σαφώς βλέπω ορισμένους κινδύνους από τους χειρισμούς ή να το θέσω διαφορετικά. Ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ήθελα την δική μας νομοδότηση να είμαστε ξεκάθαροι και αμονομικής απόψεως για να μπορούν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να το λάβουν υπόψη τους. Η ρήτρα αλληλεγγύη δεν μπορεί να ισχύσει ένα τέτοιο τομέα. Ε, και αυτό ισχύει και για αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 225 ε, και ως ε, νομική βάση. Θα πρέπει να δούμε την έννοια αυτή επί οριζοντίας βάσεως. Στο άρθρο 225 αυτό το οποίο αναφέρεται συμπεριλαμβάνει τομείς που θα πρέπει να ε, είναι ε, η αρμοδιότητα σε αυτή την ε, περίπτωση. Και λαμβάνουμε υπόψη και την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 225 μιλά και για παροχή βοήθειας και αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μιλάει συγκεκριμένα για αυτά τα οποία γίνονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από πολιτικές βλέψεις. Επομένως δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για παρεμβάσεις εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Άμυνας. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διαφωνήσω με την τροπολογία ε, ε, στο 2β για την αρχή της αλληλεγγύης γιατί εδώ υπάρχει μια σαφής ευρωπαϊκή κατεύθυνση υπό την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια νομιμοποίηση για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα λεπτό συνταγματικό σημείο και γι' αυτό, επειδή μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη, θα πρέπει η Επιτροπή μας ε, να διευκρινίσει πάρα πολύ καλά ε, το ποια είναι η ισχύουσα πρακτική μέχρι τώρα για την ε, ρήτρα αλληλεγγύης. Και η χρήση στρατιωτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 225, αυτό θα πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο και την περιγραφή, διότι ισχύουν συγκεκριμένες συνταγματικέ διατάξεις και όσον αφορά συγκεκριμένα τη Γερμανία, αυτά είναι και θέματα του εθνικού μας δικαίου και του εθνικού μας συντάγματος. Επιτρέψατε μου αγαπητοί συνάδελφοι να προσθέσω και ακόμη κάτι. Το άρθρο 225 νομίζω ότι αποτελεί ένα βασικό καθήκον, ε, περιγράφει ένα βασικό καθήκον των κρατών μελών και ο συγκεκριμένος χειρισμός για τη ρήτρα αλληλεγγύης δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς. Αργότερα ε, διευκρινίστηκε με διατάξεις του Συμβουλίου είναι κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα και ανεξάρτητα από το ε, εάν και κατά πόσο δεσμευτικά μπορεί να υπάρχουν πολιτικές ε, αναγκαιότητες και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και το 2008 είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο για το άρθρο 225 και για το θέμα της ε, πολιτικής άμυνας και των ε, φυσικών καταστροφών επίσης είχε προταθεί κάτι ε, αντίστοιχο. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει ε, να ρωτήσουμε το Συμβούλιο, θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να διεκπαιρεώσει τα δικά του καθήκοντα και να μας πει ποιοι είναι οι τομείς εφαρμογής, ποιες είναι οι αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 225 και πώς θα πρέπει να ισχύσουν ε, αυτές οι ρήτρες για τη ρήτρα αλληλεγγύης, τι όροι ε, υπάρχουν και τι συνθήκες πρέπει να πληρούνται Και Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι τη ρήτρα αλληλεγγύης τη θεωρώ ένα ε, σημαντικό εργαλείο που δεν θα πρέπει η εφαρμογή του να συνδέεται με αυτοματισμούς και με αυτόματη λειτουργία σε σχέση με ε, την ε, κάθε φορά ενδιαφερόμενη χώρα. Κατανοώ ότι πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μου πούν ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκα αυτά που λέω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό αφορά άμεσα το, τη νομική βάση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στακόφσκι έχει ξανά εγγραφεί από ό,τι βλέπω να μιλήσει. Παρακαλώ. Συνήθως είναι βαρετά αυτά που συζητάμε. Όμως είδα ότι όταν έχουμε τη live μετάδοση από το ίντερνετ, τότε ξαφνικά μυστηριωδώ γίνονται όλα ενδιαφέροντα και εγώ τέλο πάντων για τα πρακτικά, για την ιστορία έχω να σας πει ότι και εγώ είμαι κατά του να έχετε πυρηνική αποτροπή στη, στη, χώρα σα στο Μένο Βασίλειο, και, αλλά και ο κύριο Ντάφ από ό,τι ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά φιλοδοξία να γίνει αρχιστράτηγο του Ευρωπαϊκού Στρατού. Τι να σας πω. Ελπίζω να ζήσουν να το δω. Ελπίζω τώρα, τώρα να, να, να έχουμε εδώ πέρα τις, τις κάμερες να με παίρνουν εδώ ζωντανή μετάδοση και που, και που λείπει ο κύριος Αντωνότση. Τέλος πάντων, ευχαριστώ τον κύριο Άντριου που συνεφώς με τα είπα για την αδερφικότητα, για την ε, αμοιβαία ε, αρρωγή. Και υπάρχει αυτό το θέμα του Βερολίνου συν και έχουμε αυτό το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουμε επομένω όπω και τόσο καιρό επικάλυψε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το καταφέρουμε αυτό και κυρίω με τακτική, συστηματική συνεργασία μεταξύ του υπάτου εκπροσώπου, του Γενικού Γραμματεία του ΝΑΤΟ κλπ. Και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το μόνο σημείο προστριβή το οποίο απομένει σε σχέση με το Βερολίνο και βέβαια ξέρω, ξέρω γιατί γίνανε αυτά τα προβλήματα. ομω έτσι κι αλλιώ υπάρχει δεδομένη απόφαση του ΝΑΤΟ να αξιοποιήσει αυτό το σύμφωνο, ιδίως όσον αφορά τα, πρακτικά, το υλικό, ούτως υπήν, τμήμα του συμφώνου. Οπότε παρακαλώ, Άντριο, λάβε και αυτά που είπα τώρα υπόψη. Ωραία. Ο συνάδελφος Νταφ παραδόξως, ε, σήμερα το απόγευμα τελικά απεδείχθη πολύ ελκυστική αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ήταν ο αρχικός στόχος του κυρίου Πάσκου ή ο δικός μου να ξεκινήσουμε πόλεμο. αλλά να καθορίσουμε το πότε το άρθρο 42.7 μπορεί να ισχύσει, αλλά ούτε αυτό ήταν ο κύριος στόχος μας. Ο κύριος στόχος της έκθεσης ήταν να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή την, της ρήτρας αλληλεγγύης. Ο κύριος Σόλτ έχει δίκιο σε γενικές γραμμές ότι οι πολιτικές αρχές ε, του κάθε κράτους μέλους είναι αυτές οι οποίες τελικώς αποφασίζουν ε, να την χρησιμοποιήσουν ή όχι. δεν είναι δυνατόν και εμείς δεν προτιθέμεθα να επιβάλλουμε οποιαδήποτε αρρωγή, συνδρομή είτε από την Κάθη Άστον ή από τον πρόεδρο Μπαρόζο ή από τον ε, πρόεδρο Ρόμπο ή από μένα ή από οποιονδήποτε άλλον. Μπορεί κανείς να ζητήσει την ε, ενεργοποίηση της ρήτρα, ε, να δεχτεί την βοήθεια βάση της ρήτρα σε μια περίοδο κρίσης, μπορεί να κάνει όπως νομίζει. Και νομίζω ότι αυτό σαφώ ε, και ρητά το αναφέρει η έκθεση του κυρίου Πάσκου. Επομένω, κατά αυτή την έννοια, ε, δεν συμφωνώ πολύ με αυτό που ο κύριος Σόλτ, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να, ε, να βρούμε κατά αποκλειστικότητα τις αιτίες της κρίσης που θα ενεργοποιήσουν την ρήτρα αλληλεγγύης. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι στον κόσμο υπάρχουν πολλές απειλές. Η τρομοκρατική απειλή, αλλάζει μάλιστα το πρόσωπο της τρομοκρατίας ε, και οι μορφές που παίρνει είναι πολλαπλές και διαρκώς εξελισσόμενες. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να προσκοληθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη περιγραφή της ε, τρομοκρατικής απειλής. Χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας. Νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστική προσέγγιση και αυτό χρειαζόμαστε, πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Για το άρθρο 42, 7. δεν έχει γίνει καμία πρόταση να ενεργοποιηθεί ή να προχωρήσουμε περισσότερο από το πρωτογενές δίκαιο. Και πρέπει να πω στην κυρία Γιαννάκου ότι εκπλήσωμε, εκπλήσωμε από την αντίθεση της στα όσα ο κύριος Πάσκου και εγώ λέμε εδώ. Το ΝΑΤΟ ε, παρουσιάζεται στο 42 σαν ένα εργαλείο ε, κοινής άμυνας της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προσπαθούμε καθόλου να το ε, δυναμητήσουμε αυτό ή να το υποκαταστήσουμε. Δεν θέλουμε να δυναμητήσουμε, λέω, το ΝΑΤΟ, ζητώντας ή δημιουργώντας μια ε, ολοκληρωμένη στρατιωτική ευρωπαϊκή δύναμη. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Επίσης ε, είναι σαφές ότι ο βρετανικός ε, λαϊκίστικος τύπος έχει προσπαθήσει να στρεβλώσει το σημείο αυτό. Ε, το οποίο όμως καλύπτεται σαφώς από τη συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να καλλιεργούμε και να προκαλούμε φόβους χωρίς λόγο. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν αναφέρει ρητά καμία κοινή πολιτική ασφάλειας λέει ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι τέτοιες, ε, μάλλον όταν θα καλυφθούν οι πολιτικές συνθήκες, ε, τότε ε, σε κάποιες χώρες μέλη επιτρέπεται κάτι τέτοιο και η μορφή θα είναι αυτό που ονομάσαμε κοινή δομή συνεργασίας στην άμυνα. Δεν είναι αυτή όμως η εστίαση ή ο σκοπός της έκθεσης αυτής. Χαίρομαι γιατί ακούω ότι οι τροπολογίες μου έχουν ε, ενσωματωθεί στις συμβιβαστικές του κυρίου Πάσκου. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει με την ΑΦΕΤ Επομένως δεν θεωρώ ότι η Επιτροπή Συνταγματικών ε, Υποθέσεων θα πρέπει να εγκαταλείψει τις τροπολογίες αυτές ε, διότι απλά και μόνο ο εισηγητής, ο κεντρικός εισηγητής τις έχει ενσωματώσει στις δικές του συμβαστικές λύσεις. Δεν μπορώ να ακολουθήσω και να κατανοήσω τη λογική αυτής της ε, διατύπωσης που έκανε η κυρία Γιαννάκου προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει αύριο να κάνουμε την ψηφοφορία ε, και βεβαίως να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν στην συζήτηση αυτή σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία λοιπόν, συζητήσαμε αναλυτικά την, ε, έκθεση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Είμαι στο σημείο 6, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, στο πέμπτο είμαστε, ναι, ναι, στο πέμπτο σημείο της μεσής διτάξεως. Προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Συντάξει της νομοδότησης ο ε, συνάδελφος Γκουαλτιέρη. Ε, την 17η Σεπτεμβρίου στη συνεδρίασή μας του ανατέθηκε η σύνταξη της ε, γνωμοδότησης για την οποία αναρμόδια επί της ουσίας είναι η, ε, η κυρία Μαριάν Τίσεν της Οικονομικής ε, Επιτροπής. Στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφίσει η ΕΚΟΝ, άρα εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο αν θέλουμε να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση. Δεν έχουμε μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες, αλλά βεβαίως θα υπάρξει μετάφραση για την επόμενη φορά. Ο κύριος Γουαλτιέρε, αν δεν κάνω λάθος, έχει 82 τροπολογίες. Κύριε Γουαλτιέρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Τίσεν για την ίδια έκθεση έχει 950 τροπολογίες, άρα και πάλι καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους σκιώδεις ηγητές, αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους, γιατί έδειξαν πάρα πολύ καλή διάθεση επικοδομητικής συνεργασίας και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν, μας επευλήθη ένα χρονοδιάγραμμα πολύ περιοριστικό γιατί η ΕΚΟΝ ήθελε να εγκρίνει την έκθεσή της ήδη στα μέσα Οκτωβρίου ε, και μετά στην Ολομέλεια. Ε, στην πραγματικότητα, όπως είδαμε και στην τελευταία συνεδρίαση, μάλλον αυτή τη μία συνεδρίαση των ΣΕΡΠΑ την προηγούμενη, την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Δεν το λέω μόνο για εσά αλλά για όλους. Στις 5 έχουμε τους ε, ε, εισηγητέ, ε, συγγνώμη, τους συντονιστές. γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Δεν το λέω για σας κύριε Γκουαλτιέρη, μόνο το λέω για όλους. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έγινε η πολυμερή συνάντηση των ΣΕΡΠΑ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και κατέστη σαφές ότι η ενδιάμεση έκθεση του Οκτωβρίου δεν θα είναι τελειωτική και επομένως η πολλή δουλειά ε, μεταφέρθηκε για τον ε, ε, Δεκέμβριο. Όμως η έκθεση Tyson θα ψηφιστεί όπως είπατε στον Οκτώβριο, άρα πιεζόμαστε και εμείς. Ίσως και αυτό να μην είναι κακό τελικά, διότι φρονώ ε, πως ε, εκθέσεις ε, η έκθεση κύρια Τάιζεν που είναι σε πρωτοβουλία, είναι λίγο πιο περιορισμένη. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε περισσότερα πράγματα για την, στην έκθεση της διακυβέρνησης. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω για τις τροπολογίες, οι οποίες κατά την άποψή μου εμπλουτίζουν το σχέδιο γνωμοδότησης. Δεν αντιτίθενται ε, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες ε, στην ουσία της γνωμοδότησης και μου έδωσαν ε, την δυνατότητα να εκπονήσω συμβιβαστικές ε, τροπολογίες τις οποίες υπέβαλα σήμερα το απόγευμα εις τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, που νομίζω ότι καλύπτουν όλες τις προτάσεις οι οποίες υπευλήθησαν. Ιδιαιτέρως σε μια σειρά σημείων πιστεύω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες ακολουθούν και την λογική του εγγράφου των ΣΕΡΠΑ που δεν είναι επίσημο έγγραφο αλλά ε, που όμως εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη διάσκεψη των Προέδρων και ε, που με συνθετικό λοιπόν τρόπο δείχνει ε, ποιες είναι οι γενικές γραμμές της θέσης του Κοινοβουλίου. Στις συμβαστικές τροπολογίες πάντως εγώ θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω και να κάνω αναφορά στην διατύπωση του κειμένου των ΣΕΡΠΑ. Επί της ουσίας τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ε, αναθεώρησης ε, των συνθήκων, νομίζω ότι είναι ορθό ε, τουλάχιστον έτσι βλέπω στο πνεύμα των τροπολογιών των συνέλεφων Έφλερ και Ντάφ, ε, πιστεύω, λέω, ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί περαιτέρω η πρόταση που κάνουμε εμείς, η επιλογή που προτείνουμε, δηλαδή να δοθεί ε, προτεραιότητα ε, στα σταθερά στοιχεία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μεταρρύθμιση των ε, συνθήκων ε, και λαμβάνοντας υπόψη και το έγγραφο των ΣΕΡΠΑ αυτή η διατύπωση της ανάγκης οργανικής μεταρρύθμισης των συνθήκων έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι απαραίτητη. Έστω και αν ε, εγώ δεν προτίθεμαι να δεχτώ τις τροπολογίες οι οποίες θέλουν ήδη σε τούτη την έκθεση να αποσαφηνίσουν θέματα δεδομένα για ε, μια επόμενη ε, για, ένα επόμενο ε, κείμενο συνθήκων εδώ σε αυτήν την γνωμοδότηση δεν προτείνουμε συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συνθήκων προτείνουμε κατευθύνσεις Επομένως ε, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί ε, αυτή η ε, κατανόηση της ανάγκης για τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρξει λοιπόν μια ουσιαστική οργανική μεταρρύθμιση των συνθήκων. Όμως δεν θέλω εδώ να βάλουμε είτε ημερομηνίες είτε της επόμενης συνταγματικής συνθήκης, είτε ε, περιεχόμενο κτλ. Απλώς να πούμε ότι το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε θα ασκήσει εν ευθέτω χρόνο ε, ε, το, τα δικαιώματά του ε, τα δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχει όσον αφορά τις συνθήκες βάσει ακριβώς των ε, αρμοδιοτήτων που του δίνουν οι συνθήκες. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, νομίζω ότι η πρόταση του συνέλεφου Έφνερ να προτιμήσουμε την ε, δέσμη σε σχέση με τα 126.6 και 114 ε, αντί την ενεργοποίηση της ε, πασαρέλας που όμως εγώ θα την διατηρήσω σαν αναφορά ε, γιατί αναφέρεται και στο έγγραφο των ΣΕΡΠΑ αλλά θα προτιμήσω τη διατύπωση ΕΦΝΕΡ όσον αφορά την διαθεσμική διοργανική συμφωνία όσον αφορά την εξάντε, τον εξάντε συντονισμό των οικονομικών πολιτικών νομίζω ότι υπάρχει λογική στη θέση του ΕΛΚ αλλά χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για την ώρα. Να κάνουμε λοιπόν, να περιοριστούμε σε μια γενική αναφορά αυτού του ενδεχομένου. Ε, συμφωνώ λοιπόν να εγκαταλείψω ένα τμήμα του κειμένου μου ε, όπως προτείνει ο Σαρστατρακόφσκι αλλά θα ήθελα ε, να κρατήσουμε την αναφορά όπως κάνει και το κείμενο των ΣΕΡΠΑ ε, ε, στο ενδεχόμενο εξάντε συντονισμού των ε, οικονομικών πολιτικών γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι και αυτό έχει αναφερθεί και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Όσον αφορά τώρα την, την θέση από κοινού των μηχανισμών σταθερότητας νομίζω ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ότι πρόκειται για μια πρόταση η οποία θα πρέπει να μπει σε μια πιο μακρόθωρη λογική, όχι σε μια λογική άμεση υλοποίησης. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του προϋπολογισμού ε, της ε, Ευρωζώνης, ε, νομίζω ότι οι τροπολογίες του Ραφάλ Τζαρκόφσκι είναι πολύ σωστές. Η συζήτηση αυτή είναι απαραίτητη και δεν θα πρέπει να την αντιληφθούμε σαν μία ή να την εκλάβουμε σαν μία συζήτηση η οποία θα πρέπει ε, κατά κάποιο τρόπο να αποβεί προς ζημία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, γι' αυτό θα δεχτώ την ε, τροπολογία του Ραφάλ Τραυσκόβσκη για το σημείο αυτό. Όσον αφορά τα άλλα σημεία, είναι ελάσσονο σημασίας κατά την άποψή μου και ε, βεβαίως καλό θα ήταν ε, να τα ε, συζητούσαμε και αυτά στην συνάντηση των ΣΕΡΠΑ και θα ήθελα να πω και δύο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι όπως είπε και ο Πρόεδρος δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω υπερβολικά, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο διάθεση Ευχαριστώ πολύ, Σνάνφε Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε τι αποσκοπούμε και τι προσπαθούμε να ορίσουμε. Δηλαδή, μία ομοσπονδιακή οικονομική κυβέρνηση για μια δημοσιονομική ένωση. Επίσης πιστεύω ότι δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικό κοινοβούλιο πριν να έχουμε πραγματική κυβέρνηση και θα πρέπει ε, να δούμε ποια είναι η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου, σε τι βαθμό έχει φιλοδοξία το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε μια τέτοια οικονομική, πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτό πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να σεβόμεθα το διαχωρισμό των εξουσιών και θα ήταν ανόητο να προσπαθεί το Κοινοβούλιο ε, να συμμετάσχει στις αποφάσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής και του Συμβουλίου για μια κοινή δημοσιονομική πολιτική αν θέλουμε να ασκούμε και, και το καθήκον μας αυτών που κρίνουν την κυβέρνηση. Ε, και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα η έκθεση της προχωρεί υπερβολικά. Προσπαθεί νομίζω να μεγεθύνει το, το ρόλο του Κοινοβουλίου. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά το ρόλο του Προέδρου. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Δεν έχει εντολή να διαπραγματεύεται πολιτικά σχετικά με το μέλλον μιας ε, οικονομικής πολιτικής. Θα έπρεπε να του ζητείτε να συμμετάσχει και θα έπρεπε να είναι παρόν στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχόλιο προς τον κύριο Γκουαλτιέρη, ο οποίος μίλησε εκτός μικροφώνου. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε πιο αυστηρά το ρόλο του Κοινοβουλίου. Η Τρόικα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Η Τρόικα αποτελείται από την Επιτροπή που λογοδοτεί προς εμάς και προς το Συμβούλιο. Περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει διαφορετική σχέση με μας και θα πρέπει να παραμείνει η ανεξαρτησία της στα θέματα νομισματικής πολιτικής και υπάρχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Τρόικα που κατά κανένα τρόπο δεν είναι υπόλογο προς εμάς. Και αν προσπαθήσουμε να μπούμε στις εκτελεστικές αποφάσεις της Τρόικα, θα φοβούμε ότι θα δημιουργήσουμε νομικά προβλήματα. Και μπορεί να διαταράξουμε και την ηρεμία των χρηματοοικονομικών αγορών. Θα ήθελα να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο να δεσμευθεί ότι θα ζητήσει μια συνέλευση, τη σύγκληση μια συνέλευση στην άνοιξη του 2015. Γιατί νωρίτερα όλοι ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε, και όπως λέει και ο κ. Γκουαλτιέρη τελικά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη μια μεταρρύθμιση της συνθήκης και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν για να κωδικοποιήσουμε τα μέτρα διαχείρισης κρίσης τα οποία έχουν ληφθεί για να αντιμετωπίσουμε το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε. Και για να ορίσουμε πιο προσεκτικά αυτό το οποίο εγώ ανέφερα ως ομοσπονδιακή οικονομική κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει ε, να έχει και κάποιον ε, Υπουργό Οικονομικών αυτή η κυβέρνηση και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε ε, να προσδιορίζουμε τις εξουσίες του μελλοντικού Υπουργού Οικονομικών. πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ποιες θα είναι οι εξουσίες εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με αυτά που προτείνει η Επιτροπή. Διότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και αποκλείεται και ο τομέας των ασφαλιστικών εταιριών από αυτή την εποπτεία. Προτείνω τελικά να δημιουργήσουμε ε, ένα γεφύρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Αφετέρου. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αναβαθμισμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ή θα μπορούσε να είναι μια συγχώνευση των δύο εποπτικών μηχανισμών που δημιουργούμε που έχουν δημιουργηθεί από το 2008. Και θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να καλύπτει όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για το πλήρες φάσμα, για τον πλήρη τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και πιστεύω ότι στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να εκφράζουμε τέτοιες ιδέες, οι οποίες πρέπει να ακούγονται και να κυκλοφορούν στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να συζητηθούν στο πλαίσιο των επικοδομητικών συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων. E Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ και τώρα κύριος Ταρκόσκι. Πάρα πολύ σύντομα να σας μιλήσω για αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Διότι πρόκειται έτσι καλώς να τα συζητήσουμε για το ευρύτερο θέμα στο μέλλον. Και εδώ δικαιούνται πάρα πολλά, οι υπόσχεσεις με τι αμμουδιότητες σε σχέση με την Τρόικα, σε σχέση με του Σέρπα και πάντω όσον αφορά αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ρομπέρτο, διότι ο Ρομπέρτο έλαβε υπόψη τα περισσότερα από τα αιτήματά μου στι τροπολογίε και νομίζω ότι αυτό που θέλεις να μιλήσεις για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμη σαφήνεια στο έγγραφο μας ε, έδωσες μια αφορμή να προχωρήσουμε, να δουλέψουμε και να έχει έτσι ουσιαστικό περιεχόμενο αυτός ο γιατί πρόκειται για εξελίξεις για το μέλλον δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ευθύς αμέσω και ξέρεις ότι αυτό που με προβληματίζει κυρίω είναι ότι ό,τι και να κάνουμε Ε, αυτά που θα αποφασίσουμε για τα φορολογικά θα έχουν άμεση επίπτωση στην επεξεργασία του σχεδίου προπολογισμού. Άρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτές με τις θέσεις σε σχέση με τι θα γίνει μέσα στον, δια, στον προπολογισμό και ταυτόχρονα να μην υποσκάψουμε ε, τις πολιτικές που χαράσουν επί τη βάση του προπολογισμού. Αυτό με απασχολεί επίση, Άντριο είναι κάτι που συνδέεται με το επόμενό μας θέμα γιατί θα ασχοληθούμε και με τον προπολογισμό με άλλη μια έκθεση. Αυτά τα οποία βρίσκονται τώρα επί τραπέζης θα πρέπει να μας αποσχολήσουν όσο γίνεται πιο σοβαρά. Να κλείσουμε συμφωνία για τον προπολογισμό εν του 2020 πρώτα και κατόπιν να δούμε πώς θα σώσουμε την ε, implications in our future debate, uh, such as questions such as creating this new capacity, such as questions of. Πέρα από την νομισματική ένωση. Και έτσι να δούμε το ότι ο μηχανισμός στήριξης είναι η πιο σωστή προσέγγιση. Επομένως, έχουμε με δεδομένο το χρονοδιάγραμμα αυτό και άρα έχουμε και τη σωστή στρατηγική να συζητήσουμε και στα δύο μέτωπα. Να τα συζητήσουμε βέβαια παράλληλα και ξεχωριστά όσο γίνεται παρά το ότι αλληλοσυνδέονται. Όμως εάν δεν λυθεί το θέμα του προεμπορισμου 2014 2014-2020 και μετά να δούμε πώς θα σώσουμε την ομισματική Ένωση, τότε θα υποσκάψουμε την θέση, τη φωνή του Κοινοβουλίου, αλλά είμαστε φιλόδοξοι, θα προωθήσουμε και τα δύο θέματα και γι' αυτό το λόγο καλύτερα να μείνουμε πιστοί σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και επίσης να είμαστε όσο γίνεται πιο σαφείς. Όπως είμαστε και τώρα για αυτές τις σημαντικές τοπολογίες, για να δούμε τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι διαπραγματεύσει θα γίνουν σε ποια σημεία. Υπάρχουν πάντως ε, πέραν ε, των όσων ε, είπες για τον Τάισιν και για τη μεθοδολογία. Έχω να πω το εξής. Εγώ δεν θέλω να δυναμητήσω την διαδικασία αλλά να έχουμε υπόψη το τι πρεσβεύουν συνάδελφοι σε άλλες επιτροπές και ποια είναι η τελική θέση του Κοινοβουλίου. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικής δουλειάς και προσεκτική ταυτόχρονα στο τι θα συζητηθεί, τι θα γίνει στο μέλλον ούτως ώστε να μην είναι αυτοκτονικό, μην, μην προσκάψουμε οι ίδιοι τη δική μας θέση. Προσπαθώ δηλαδή να σας πω ότι υπάρχουν ε, ε, διαμαρτυρίες, υπάρχει γκρίνια ακόμη στη δική μου πολιτική ομάδα. Προσοχή, μην κάνουμε πράγματα αντιπαραγωγικά, ακόμα και αν ε, υπάρχει σε τεχνοκρατικό επίπεδο συμβιβασμό. δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε συνολικό συμβιβασμό, το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε μήπως οι ίδιοι αργότερα το ανατρέψουμε. Αυτό επισυνδέεται με κάποια προβλήματα το οποίο ποτέ συνδέονται στο Κοινοβούλιο. For Την έκθεση επομένω, έχω πει ότι αν προχωρήσουμε τι διαπραγματεύσει, αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν. Όμω, πολλέ φορέ με την εντύπωση ότι κάποια θέματα, όπω αυτό για την Τρόικα Φερρυπίν, πάνε πέρα από αυτά. Και αν δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών για αυτές τις συζητήσεις. Με, τους συνήθιους τρόπους και διαδικασίες τότε ίσως αυτό σημαίνει ότι θα βλάψουμε τους εαυτούς μας. Αυτό όσον αφορά την γνωμοδότηση είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με αυτό το οποίο είπες με τη βάση των συζητήσεων των επαφών, το έγγραφό σας που έγινε βγήκε μετά συνήθως με τους άλλους Σέρπα και πάλι σας ευχαριστώ. Κολέγα Μπρόντς, αλλά παρόλα. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρόντς. Χωρίς μικρόφωνο. Η Βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό το θέμα είναι τελείω άσχετο με χώρε εκτό Ευρωζώνη και είναι τελείω άσχετο με το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει αυτό εξαιρεθεί. Όμω, τον Δεκέμβριο τουλάχιστον ε, δείξατε μία μικρή, μία μικρή αντικρότηση. να μην επιβάλλετε σε όλου αυτό που θέλετε να κάνετε στον εαυτό σας. Εμείς πάντως αυτό το οποίο πρεσβεύουμε σημαίνει ότι δεν θέλουμε με τίποτα να έχουμε αυτό το ζωολομανδία ε, και, και, να, για να μα δέστε χειροπόδαρα όλους με, με την Ευρωζώνη, γιατί το ε, σύμφωνο αυτό δεν ισχύει για μας. Άμα κάποιο βέβαια θέλει μόνος του να δεσμευτεί σε μια κατάσταση, δεν πρέπει να παραπονιέται μετά. Όπω ε, ό,τι βγήκε για, ε, στο Δημοσίου τη Λισαβόνα, θα βγει και τώρα, άμα γίνει δημοψήφισμα. Και από ό,τι λέει ο εισηγητή, η εποπτεία και ο δημοσιονομικό ένωμο των χωρών τη Ευρωζώνη θα μπορούσε να γίνει δεσμευτικό και να επιδέχεται και δικαστικό έλεγχο από το ΔΕΚ εάν το άρθρο 136 τροποποιηθεί τη Συνδική την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παραγράφος 6. Και μετά μας είπατε ότι θα πρέπει αυτά να τα επικαλούμεθα μόνο εάν ενισχύει το ρόλο του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ε, ε, ερμηνεία αυτών των δύο άρθρων. Παρακαλώ αν μπορείς εξήγησε με αυτό και δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ τον κύριο Γκαλτιέρη, γιατί χωρί να ρωτήσω, χωρί να διαβάσω τι λεπτομέρειε των όσων είπε, ε, δεν ξέρω τι θα γίνει το άρθρο 121 αυτή τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι ακριβώς εδώ που θα διάβαζα πριν πέσω να κοιμηθώ. Όμως η διαδικασία του 120 λέει ότι τα κράτη-μέλη πρόκειται να ασκούν την οικονομική του πολιτική εν ώψη του να επιτύχουν του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο άρθρο 121 μετά στη συνέχεια ορίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επαναχαράξουν τις εθνικές πολιτικές σαν, σαν ε, ένα θέμα κοινής μέρημνας και να συντονιστούν μέσω του Συμβουλίου σύμφωνα με το όσο ορίζει το άρθρο 120 και παρακάτω έχουμε το 121.4 το οποίο αναφέρει ότι ορίζεται ότι δεν θα πρέπει οι των μελών να θέτουν κινδύνο τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο μπορεί να δυνατόν να απευθύνει μια προειδοποίηση η Κομισιόν ή στα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα από αυτά, λένε το 121, δεν κάνουν διάκριση όσον αφορά αυτέ τι χώρε εντό και εκτός της Ευρωζώνης. Όμως εδώ πέρα αυτό το χωρίο εμφανίζεται ως απόκληση από, το, από παράγραφο 1 παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Τα ξέρω αυτό και διάβασα το βιβλίο του κ. Ντάφ. Ε, βέβαια όλα αυτά μεταφέρουν διάφορους τρόπους στο λαϊκό τύπο, αλλά όταν θέλετε να διαβάσετε το νομοθέτημα όσον αφορά σημαίνει ότι αυτές, αυτοί οι περιορισμοί που τώρα επιβάλλονται στην Ευρωζώνη θα μπορούσαν με κάποιες μικρές αλλαγές να επιβληθούν και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Βεβαίω θα πρέπει κανείς να περιμένει και να δει κάτι Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη για την τελική του απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay, start to reply to some of the points. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε ορισμένα από τα σημεία που ανέφεραν οι συναδελφοί μου. Πρώτον, τα σχόλια του κύριου Ντάφ. Σχετικά με, το, με την Προεδρία δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα του Κοινοβουλίου Υπάρχει μια παράγραφος της εκθέσεως της κυρίας Τάισεν σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαβουλεύσεις για την ε, προετοιμασία της έκθεσης. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και, και θα υπάρχει και μία νέα εκδοχή πιο επικαιροποιημένη, αλλά η πρότασή μου είναι να παραμείνουμε σε γενικές γραμμές και απλώς να λάβω με γνώση των όσων έχουν ε, συμβεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον... Εμ, ενσωματωθεί στη διαδικασία και έχει στείλει κάποιους σέρπας. Αλλά νομίζω, και αυτό είναι σημαντικό ε, να αποσαφινιστεί, ε, για, κυρίως σε σχέση με τα πολύ σημαντικά σημεία που ανέφερε ο συνάδελφος ε, Ράφελ Ταρκόφσκι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Ε, η, εργασία του Κοινοβουλίου είναι, συν, είναι εργασία συνσυντάκτου κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε ακριβώς έτσι για την έκθεση Φαν Ρόμποϊ. Ε, υπάρχει απόφαση για διαβούλευση. Νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κρατήσει την δικιά του θεσμική αυτονομία ε, για θεσμική και συνταγματική πρωτοβουλία που είναι ξεχωριστό από το ότι είναι μέρος μιας διαβουλευτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στην έκθεση Βαν Ρομπόη και όχι στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι σαν Κοινοβούλιο έχουμε το δικαίωμα να ε, ζητήσουμε τη σύγκληση ε, συνθήκης ε, ε, και χρησιμοποιούμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι η διατύπωση που προτείνω εγώ, δηλαδή γνωρίζουμε, συνειδητοποιούμε την ε, δυνατότητα πρωτοβουλίας που έχουμε και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, είναι καλύτερη διατύπωση. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, άποψή μου και με αυτό απαντάω και στο σημαντικό σημείο που έφτιαξε ο Ράφε και στην έκθεση Tyson και ε, στην ε, έκθεση ε, Σέρπα δεν υπάρχει πρόθεση να μπούμε σε νομοθετική διαδικασία εμείς εμείς έχουμε επανειλημμένα ε, αναφέρει την πρωτοκαθεδρία της ε, κοινοτικής διαδικασίας και τώρα στον εποπτικό μηχανισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα, ε, μια έκθεση σαν της κυρίας Τάισεν ή ακόμα χειρότερα μια μια ε, έκθεση σαν αυτήν τον ΣΕΡΠΑ ε, και να την αναμίξουμε με την νομοθετική πρόταση. Και στο έγγραφο ΣΕΡΠΑ βλέπουμε ότι η αστίαση γίνεται σε γενικό τεχνικά ζητήματα μεθοδολογίας και γενικά συνταγματικά ζητήματα. Δεν μπαίνει σε ε, λεπτομέρειες νομοθεσίας. Σε γενικές γραμμές πάντως συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο Ταρκόφσκι και τις ε, ε, σχετικά με την ανάγκη να μην αγνοήσουμε βεβαίως θέσεις και ευαισθησίες και ε, ε, συζητήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει ε, στις επιτροπές και στις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό ο, λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς δεν θα είμαστε συν αλλά γίνεται διαβούλευση και με μας ε, και εμείς χρησιμοποιούμε την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε θεσμικά ζητήματα. Πρώτον, ότι δεν θέλουμε κανένα διαχωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις τρεις αρχές ε, που αναφέρονται άλλωστε και στο έγγραφο ΣΕΡΠΑ, που είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να το έχει κανείς στην ε, έκθεση Tyson. σχετικά με την Τρόικα. Αυτό που προτείναμε σε κάποιες τροπολογίες αλλά και στο έγγραφο ΣΕΡΠΑ είναι να μην μπερδεύουμε τον ρόλο ε, του, εκτελεστικού οργάνου και ε, του ε, ελέγχου. Απλώς θα πρέπει να καταδειχθεί η δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικα που αυτή τη στιγμή υπολείπεται. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει. Αυτό το σώμα έχει ε, σημαντικές ε, δικαιοδοσίες και βεβαίως θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα ε, στον εκτελεστή, στην εκτελεστή λειτουργία και τον έλεγχο, το θεσμικό έλεγχο και βεβαίως όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της σωστής δημοκρατικής λειτουργίας. Και αυτό αναφέρεται άλλωστε και σε κάποια σημεία του εγγράφου των ΣΕΡΠΑ και νομίζω ότι και η ίδια η κυρία Τάισεν θέλει να ενσωματώσει το σημείο αυτό της Τρόικας στην έκθεσή της. I don't uh, Δεν ξέρω αν έχω τίποτα άλλο να πω τουλάχιστον όσον αφορά το μέσο ή μακροπρόθεσμα. Στι τελευταίε ερωτήσει η απάντηση είναι πάρα πολύ ε, απλή. Έχουμε το άρθρο 136 που είναι ε, άρθρο το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για τις χώρες Ευρωζώνης. Και με το άρθρο 136 ε, σε συνδυασμό και με την ε, αντίστοιχη ε, θέση 122 είναι σαφές ότι αναφερόμαστε μονάχα στις χώρες της Ευρωζώνης. Η, αναφορά, η αναφορά που έκανα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι τεχνική αναφορά. Δεν στηρίζω δεν υποστηρίζω περαιτέρω ενδυνάμιση των μέτρων όσον αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία γιατί θα ήταν δύσκολο, θα ήταν περίεργο να ξεκινήσουμε έτσι μια νέα ε, νομοθετική διαδικασία όταν ακόμα δεν έχουμε ε, επιβάλει το Fiscal Compact και έχουμε ε, και το Tupac το οποίο ακόμα πρέπει να εγκριθεί. Βεβαίως όμως πρέπει να γνωρίζουμε γιατί βεβαίως αυτό συζητήθηκε και εδώ αναφέρω εγώ την δικιά μου αξιολόγηση, η ειδική νομοθεσία για τις χώρες ε, της Ευρωζώνης και όσον αφορά την εξάντε, ε, τον εξάντε έλεγχο, ναι αυτό θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και από το ε, δικαστήριο γιατί βεβαίως αυτό θα ήταν κάτι ξέχωρο από την γενική νομοθεσία που αφορά όλες τις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να είναι πιο σαφές τώρα. Τελευταία παρατήρηση για τον Άντριου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε μόνο για δημοσιονομική ένωση, fiscal union γιατί αυτή είναι μόνο μία διάσταση. Θα πρέπει να μιλάμε για οικονομική ένωση, για πολιτική ένωση, για δημοσιονομική ένωση και για τραπεζική ένωση έτσι ώστε να έχουμε διευρυμένη ε, έτσι, άποψη. Αλλά βεβαίως ε, συμφωνώ ότι μια ε, πλήρης οικονομική και δημοσιονομική ένωση θα απαιτήσει... Ε, θα απαιτούσε και ε, και κοινό Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Πολύ ωραία. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το σημείο αυτό. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία επ' αυτού. Έχουμε ακόμα δύο σημεία να εξετάσουμε πριν από την συνάντηση των συντονιστών. Σημείο 6. Ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Και έχουμε και το σημείο 7. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγητής ε, στο πρώτο σημείο είναι η ο κύριος Ραφάλ Ταρκόφσκι και στο δεύτερο η κυρία Ανέλη Γιάντεν δεν έχουμε χρόνο για κανονική συζήτηση τώρα, να, γιατί έχουμε τους συντονιστές, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, στο πρώτο σημείο, κύριε Ταρκόφσκι, παρακαλώ να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά την κατάσταση της γνωμοδότησης. Πάρα πολύ σύντομα. Εξέτασα ε, την ε, διάμεση έκθεση από θεσμικής πλευράς και προτίμησα να επικεντρώσω την προσοχή μου στα δύο πιο σημαντικά σημεία. Το ένα είναι η περίοδος του πολιτούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και λέγω ότι η επταετής περίοδος φαίνεται ότι είναι σωστή, ιδίω όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα και τη συνέχεια των επενδύσεων και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στην επταετή διάρκεια, ιδίω σε περίοδους κρίσης. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει τον αριθμό 5 ή 7, αλλά νομίζω τώρα είναι 7 και δεν θα πρέπει να προδικάσουμε το τι θα ακολουθήσει μετά το 2020. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Υπάρχουν αρκετές ε, ιδέες οι οποίες κυκλοφορούν και εγώ αποφάσισα να τονίσω ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει ε, ε, τα κονδύλια που δίδονται για να μην επηρεάζονται οι προσδοκίες των δικαιούχων και ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των επενδύσεων, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε περίοδους κρίσης. Και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό ως μοχλό της ανάπτυξης, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο σήμερα, δεν πρέπει ε, να δώσουμε διφορούμενα μηνύματα. Πρέπει να πάρουμε ξεκαθαρή θέση για αυτά τα δύο σημεία. Ε, τρίτον, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες παραλήψεις στις πολιτικές προτεραιότητες και γι' αυτό εγώ αναφέρω το θέμα της γειτονίας και δέχθηκα και την πρόταση του Άντριου ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε ευρύτερα, να μιλάμε για τις διεθνείς ε, ευθύνες ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησα δηλαδή να πάρω και την πρόταση του Άντριου και να τη συνδυάσω με τη δική μου για να εκφράσω τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες που θεωρώ πιο σημαντικές. Διάβασα και όλες τις δικές σας τροπολογίες ε, με μεγάλη προσοχή και προσπάθησα να δεχθώ όσες τροπολογίες μπορούσα αν και κάπου δυσκολεύτηκα σε ένα σημείο παραδείγματος χάρη για την αύξηση των ορίων του προϋπολογισμού θα μπορούσα να το δεχτώ αλλά δεν νομίζω ότι θα είχαμε συμφωνία ούτε μέσα στις πολιτικές μας ομάδες. δεν θα το πρότεινα εγώ μέσα στην πολιτική μου ομάδα κάτι τέτοιο, ακόμη και αν θα ήθελα να δεχθώ αυτή την τροπολογία. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Απλώς εγώ ήθελα να εξηγήσω γιατί προτείνω να ψηφίσουμε αρνητικά, να καταψηφίσουμε την τροπολογία του Άντριου για την σύνδεση μεταξύ της βαθύτερης, της βαθύτερης ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να τα βάλουμε μαζί. Ε, ξέρω ότι κάτι διαφορετικό εννοούσε, αλλά αν τα βάλουμε μαζί σε μία πρόταση, όπω είναι στην τροπολογία σου, θα δώσουμε λάθο εντύπωση ότι δεν συμφωνούμε ω κοινοβούλιο με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αλλά μια και μου είπατε να είμαι σύντομο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Αν και έχω κανένα δυο πραγματάκια που θα ήθελα να αναφέρω. Τέλο πάντων, αυτή είναι η θέση του εισηγητού σα για την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Σέρβο Άγνιου έχει διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να συζητήσουμε σήμερα τα σημεία 6 και 7 στην ημερήσια διάταξη. Γιατί να μην τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αν δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα. Μα έχουμε ήδη καθορίσει αύριο την ψηφοφορία επί των θεμάτων αυτών. Ή θα πρέπει να αναβάλουμε τις ε, ψηφοφορίες ή θα αρκεστούμε ε, σε μια συνθετική παρουσίαση από πλευράς των εισηγητών. Δεν βλέπω την κυρία Γιατερμάκη βέβαια. Ίσως το σημείο αυτά δεν μπορούμε καν να το συζητήσουμε. Να το αναφέρουμε καν. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το πρόγραμμα των ψηφοφοριών θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό. Πάντως αν θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση ε, στο σημείο, για το σημείο 6, επί του οποίου ήδη μίλησε ο συντάκτης ομοδότης ο κύριος ε, ε, Τσαρκόφσκι, έχουμε λίγο χρόνο. Μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε. Πολύ καλά, Πρόεδρε. Μόνο πέντε θέσει θα σα πω. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο σημεία όσον αφορά το, το, το, τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει με, τα, με, τους, με τον περιουσία των χωρών. Τι θα γίνει με αυτή την ευξημένη εργασία όσον αφορά την φορολογία, διότι τελικά αυτό είναι ε, μα, ε, μας γιατί αν κάνετε κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργήσει η δημοσιονομική πολιτική με, με αυτή τη φορολογική που θέλει να ακολουθήσετε γιατί τότε καμία χώρα δεν θα μπορεί να βάλει του δικού φορολογικού συντελεστέ και οπότε έτσι δεν θα υπάρχει κανένας είδου φορολογικό ανταγωνισμός η εναρμόνιση δεν πρόκειται να είναι κάτι που θα γίνει με συνένεση αλλά θα επιβληθεί τα κράτη με εκείνα τα οποία έχουν χαμηλού συντελεστέ, ε, ε, εκείνα τα οποία δεν θα δείξουν 100% αλληλεγγύη πρόκειται να διαταχθούν να αυξήσουν του συντελεστέ, όπω ο εταιρικό χώρο στην Ιρλανδία ήδη θα γίνει αντικείμενο τέτοια διαταγή, θα, θέλουν, θα τους πούνε να αυξήσουν και αυτό είναι η φορολογική πολιτική είναι κλασική αρμοδιότητα κοινοβουλίων και εθνικών κυβερνήσεων όταν όμως δεν μπορούν να έχουν την τελευταία κουβέντα ποια θα είναι η φορολογική πολιτική τότε η, ε, η ύπαρξη ενός τέτοιου κράτους Ετίθεται ένα αμφιβόλο. Οπότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα τα οποία τα υφαρπάζει η ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ε, αρχίσουν ε, αυτή τη διαδρομή δεν μπορούν να συστηματίσουν ποτέ οι αυτοί οι παράγοντε τη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τότε τι επόμενε εκλογέ θα απαντήσουν σωστά οι ψηφοφόροι και σε Ελλάδα και Ιταλία θα, έχουμε τεχνολογιά στην κυβέρνηση, αυτό θα θεσμοθετηθεί και τα ανεξάρτητα κράτη τα οποία τα οποία έχουν ανεξάρτητη φορολογική πολιτική και προπολογισμό. Ε, αυτά θα ανοίγουν στο παρελθόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν όλα το γεγονός ότι οι αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές έχουν ήδη ορίσει ε, ημερομηνίες ε, μας ε, περιορίζει και δικιά μας, στις δικές μας κινήσεις. Δηλαδή ή θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο ή θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως και να χάσουμε τις ευκαιρίες. Ε, κώδικας διοικητικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το σημείο 7. Δεν δεν έχουμε εδώ την εισηγήτρια, επομένω, δεν, υπάρχει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Να σα πω πάντως ότι η ψηφοφορία και για το θέμα αυτό, δηλαδή τον κώδικα διοικητική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο συντάκτια γνωμοδότηση είναι η κυρία Γιάτερ Μάκη ε, και που συζητήθηκε ήδη η γνωμοδότηση στις 29 Μαΐου ε, θα ψηφιστεί αύριο. Θα συναντηθούμε λοιπόν σε λίγο στη συνάντηση, στην συνεδρία συγγνώμη των συντονιστών.